η συζήτηση, τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση, έληξε εδώ. Και ερχόμαστε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που είναι προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή με θέμα παραπλανητικές πρακτικές των εταιριών έκδοσης καταλόγων επιχειρήσεων. Ξεκινάμε με τις παρεμβάσεις των συντακτών. Ο κύριος Μπουζουτήλ για δυόμιση λεπτά πρώτος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, πριν από δυόμιση χρόνια υπέβαλα στην ε, Ολομέλεια μια έκθεση σχετικά με τις ε, παραπλανητικές ε, επιχειρηματικές πρακτικές και το μήνυμα που έδωσε το Κοινοβούλιο ήταν σαφές. Δηλαδή ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με παραπλανητικές επιχειρηματικές πρακτικές και ότι δεκάδες και εκατοντάδες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ακόμα και φιλανθρωπικές οργανώσεις, τελικά πέφτουν θύματα αυτών των παραπλανητικών πρακτικών και ότι χρειάζεται κοινή αντιμετώπιση έτσι ώστε μία και καλή να σταματήσουν αυτές οι παραπλανητικές πρακτικές. Δυστυχώς, δυόμιση χρόνια μετά, να είμαστε πάλι εδώ να συζητούμε το ίδιο ακριβώς θέμα διότι υπήρξε σοβαρότατη έλλειψη αντιμετώπισης σωστής του προβλήματος αυτού. Και αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Να υπενθυμίσω στους συναδέλφους γιατί μιλάμε. Στην ουσία ε, μιλάμε για παραπλανητικές ε, εκδόσεις από εταιρείε έκδοσης καταλόγων επιχειρήσεων που ε, ζητούν από ε, συγκεκριμένους ε, που, από επιχειρήσεις οι οποίες ζητούν ε, να εγγραφούν στους καταλόγους αυτούς. Αυτές οι εταιρείες λοιπόν τους λένε ότι θα τους καταγράψουν δωρεάν σε αυτούς τους καταλόγους εάν δεχτούν να αναβαθμίσουν κάποιες υπηρεσίες. Και τελικά δεν γίνεται τίποτα από αυτό και στην ουσία πληρώνουν χωρίς να δέχονται καμία, ε, ε, καμία υπηρεσία. Ε, στην ουσία εδώ μιλάμε για πολύ επιθετικές πρακτικές, δηλαδή σε περίπτωση μη καταβολής των χρημάτων υπάρχει μια διαρκής πίεση μέσω τηλεφώνων, μέσω απειλών για δίθεν δικαστικές διαδικασίες κτλ και ε, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι εθνικές αρχές αυτές τις καταχραστικές πρακτικές αλλά δεν αναλαμβάνουν ε, τίποτα, δεν αναλαμβάνουν καμία δράση. Ε, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι κατάλογοι. Πρόκειται για τηλεφωνικούς καταλόγους, για καταλόγους εκθέσεων, για καταλόγους ειδικών θεμάτων που εξακολουθούν και λειτουργούν κανονικά. Μα αυτές είναι εξαιρετικά καταχραστικές και παραπλανητικές πρακτικές οποίες λειτουργούν κατά του και παρά τον Ευρωπαϊκό Νόμο. Πρέπει να σταματήσουν. Άλλη συντάκτης, η κυρία Κορχόλα, για δυόμιση λεπτά επίση. Uh, dear President, dear members. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη Αυτές οι εταιρείε έκδοσης καταλόγων επιχειρήσεων προχωρούν σε παραπλανητικές επιχειρηματικές πρακτικές και αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Ε, ε, οι εταιρείε αυτές προκαλούν πολύ μεγάλο οικονομικό βάρος, ακόμα και καταστροφή στις χώρες αυτές, συγγνώμη, στις εταιρείε οι οποίες έχουν προστρέξει τις υπηρεσίες τους. Ε, είχαμε 14.000 προσφυγές μόνο την προηγούμενη χρονιά και κάθε χρόνο έχουμε τέτοιου είδους ανα ε, νομίζουμε ότι αυτού του είδου οι πρακτικέ τέτοιων εταιριών ε, δυναμητίζουν τα ίδια τα θεμέλια τη εσωτερική αγορά. Υπάρχει ε, συγκεκριμένη οδηγία σχετικά με τις παράνομε και παρανομικές πρακτικές και αυτέ οι πρακτικέ των εν εταιριών έκδοση καταλόγων σαφέστατα εμπίπτουν στην οδηγία αυτή οι Ολλανδικές ε, αρχές ε, πρόσφατα ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό ε, και σχετικά με μια εταιρεία έκδοση καταλόγων με έδρα την Ολλανδία. Σαφέστατα καταδεικνύεται ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη ασχολούνται μόνο με όσα συμβαίνουν στην δικιά τους επικράτεια. Όμως σε διασυνοριακό επίπεδο θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία έτσι ώστε να σταματήσουν οι παραπλανητικές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση θα πρέπει να αναλάβει πιο ενεργητικό ρόλο όσον αφορά την ενδυνάμωση τη ε, μεταφορά του ευρωπαϊκού, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με όλα τα εργαλεία τα οποία ήδη υπάρχουν στη διάθεσή του. και επίση θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικέ κυρώσει για αυτού του είδους παραπλανητικέ πρακτικέ σε όλε τι ε, ε, χώρε, έτσι ώστε οι εταιρείε έκδοση καταλόγων και να φύγουν από την αγορά και να υποστούν κυρώσει. Πρόκειται για αθέμητες πρακτικές, οι οποίες, εμπορικές πρακτικές, οι οποίες εμπίπτουν στην σχετική ε, οδηγία. Και επομένως πρόκειται επίσης για πρακτικές οι οποίες ε, ε, δημιουργούν πρόβλημα στην εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στον καταναλωτή και τον επιχειρηματία. Αθέμητες πρακτικές θα πρέπει να καλύπτονται από τις ίδιες πρακτικές, αθέμητες δηλαδή πρακτικές απέναντι σε επιχειρήσεις θα πρέπει να καλύπτονται από την ίδια νομοθεσία που καλύπτει τις αθέμητε πρακτικές επιχειρήσεων ε, κατά των καταναλωτών. Θα πρέπει επίσης να βελτιωθεί ο κανονισμός και η δυνατότητα συλλογικής προσφυγής, ε, διότι διαφορετικά ε, δεν είναι δυνατόν ε, να προχωρήσουμε σε κανονική διασυνοριακή συνεργασία έτσι ώστε να μπορέσει να τελειώσει αυτό το ζήτημα με τις εταιρείες έκδοσης καταλόγων. έχει το λόγο τώρα. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται τι ανησυχίε και την ε, κριτική την οποία ασκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν ε, παραπλανητικές ε, πρακτικές από εταιρείες έκδοσης καταλόγων επιχειρήσεων και διάφορες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα λόγω αυτών των πρακτικών. Πριν από τρία χρόνια ζητήσατε να διεξαχθεί μια τέτοια μελέτη και λάβουμε πάρα πολλές πληροφορίες και θεωρούμε ότι παρόλα αυτά έχουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Δηλαδή ότι ο ρυθμός των ατόμων τα οποία θεωρούν ότι αποτελούν θύματα παραπλάνησης είναι πολλαπλάσιος. Η συνάδελφος Ρέντινγκ εξετάζει τα δικά της ε, στοιχεία επί του παρόντος για να διαπιστώσει τη διάσταση του προβλήματος καταρχάς. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι πρακτικές αυτές ε, αντιμετωπίζονται από την Οδηγία 114 του 2006 που αφορά τις ε, παραπλανητικές ε, πρακτικές στην διαφήμιση. Και ότι απαγορεύονται οι πρακτικές αυτές λόγω της νομοθεσίας πολλών κρατών μελών, αλλά διάφορες παραπλανητικές πρακτικές είναι υπερεθνικές και έτσι δύσκολα, είναι δύσκολο να καταδικαστούν. Επί του παρόντος, η συνάδελφος Ρέντινγκ σκοπεύει να καταπολεμήσει το πρόβλημα αυτό. σκοπεύει να προβεί σε ανακοίνωση στα τέλη του χρόνου σε ό,τι αφορά την οδηγία για την παραπλανητική και συγκριτική ε, διαφήμιση και να διαρευνήσει περαιτέρω δυνατότητες για την αξιολόγηση των πρακτικών αυτών. Θα προτείνει βελτιώσεις επί του περιεχομένου, συμπεράσματα από τις ε, παραπλανητικές πρακτικές που υφίστανται και θεωρεί ότι η συνεργασία με τις εθνικές αρχές σε ό,τι αφορά την ποινική δίωξη υπερεθνικών ε, περιπτώσεων θα πρέπει και μπορεί να βελτιωθεί. Επίσης ε, θα προτείνει να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ως προς τις πρακτικές αυτές και να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιότητα γενικά. Η οδηγία του 2006 έχει εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Παρ' όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν ώψη και της μελλοντική αυτής ανακοίνωσης, ζητάει από τα κράτη-μέλη να αναφέρουν τα σχετικά μέτρα που λαμβάνουν διεξάχθηκε στα τέλη ε, Μαΐου μια, ένα συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα κράτη-μέλη για να συζητηθούν τέτοια θέματα και σημείο έμφασης ήταν ακριβώς αυτές οι παραπλανητικές πρακτικές εταιριών έκδοσης καταλόγων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε ό,τι φορά διασυνοριακές τέτοιες συναλλαγές και χρειάζεται συστηματικά καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών, κρατών, ε, ε, εθνικών αρχών και η ανακοίνωση της συναδελφού Ρέντινγκ ακριβώς αυτό το σκοπό θα εξυπηρετήσει στα τέλη του χρόνου. Επειδή το θέμα είναι κατεπήγον, ε, αντιμετωπίζεται και με κατεπήγουσα τη δικασία από εμάς. Θέλουμε να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί φυσικά και η άποψη των θυμάτων, αλλά χρειαζόμαστε και κάποιο χρόνο από τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων και μετά από τον έλεγχο όλων των επιχειρημάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει περαιτέρω μέτρα για την πρόληψη τέτοιων ε, διασυνοριακών παραπλανητικών πρακτικών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έντονη υποστήριξή σα στο θέμα αυτό. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόμαστε τώρα στου ομιλητέ εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων. Έχουμε ήδη καθυστέρηση στην ε, ερωή τη ημερήσια διάταξη. Θα κρατήσετε το χρόνο σα παρακαλώ που έχει εγκριθεί για την παρέμβασή σα, και αλλιώς θα αναγκαστώ να σα διακόπτω. Πρέπει να προχωρήσουμε στι ψηφοφορίε, και μετά όπως σα είπα είναι μέρα αναχώρηση συναδέλφων. Ε, ο κύριος Παπα-Νικολάου εξ ονόματος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. 1,5 λεπτό κύριε Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι κύριε Επίτροπε δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει με τόσα είπατε. Εγώ θα περιγράψω την ταλαιπωρία που υπέστη Έλληνα συμπολίτη μου, ο οποίος μου κατήγγειλε μια αντίστοιχη περιπέτεια που είχε από τέτοια παραπλανητική διαφήμιση και μου παρέδωσε και όλα τα σχετικά έγγραφα. Έχουμε λοιπόν το έγγραφο που αποστέλει η εταιρεία αυτή που παραπλανεί η οποία ψηλά ψηλά στο έγγραφο αναγράφει ότι το updating η ενημέρωση δηλαδή is free of charge. Αυτό λέει το έγγραφο αυτό. Και ο συμπολίτης μας προφανώς βλέποντας μετά ότι πρέπει να συμπληρώσει κάποια στοιχεία συμπληρώνει τα στοιχεία και αποστέλει αυτή την επιστολή. Με πολύ μικρά γραμματάκια στο κάτω μέρος του εγγράφου αναγράφεται ότι πρέπει να πληρώνει όπως είπε και ο κύριος μπουζουτήλ προηγουμένως 1000 ευρώ το χρόνο. Ε, στη συνέχεια και αφού περνάει ε, χρόνος αποστέλει το νομικό δίθεν τμήμα της εταιρείας επιστολές έχω εδώ και τις επιστολές με την οποία από το συμπολίτη μου ζητάει 3.529 ευρώ ε, ε, ε, να καταβάλει διότι υπάρχουν και οι τόκοι και η αμοιβή της νομικής ε, συμπαράστασης της εταιρείας. κύριε επίτροπε είναι δεδομένο ότι υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο δεν ξέρουμε όμως κατά πόσο αυτές οι οδηγίες ε, εφαρμόζονται έχουν ενσωματωθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη. το πρόγραμμα της στοκχόλμης αναγράφει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα τα θέματα αυτά. είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας είμαστε κοντά και στα καθημερινά τους προβλήματα πρέπει οι, πολίτες μας, οι συμπολίτες μας να καταλάβουν δεν είμαστε κάπου μακριά δεν ασχολούμαστε μόνο με τα μεγάλα ευρωπαϊκά θέματα είμαστε κοντά τους στην καθημερινή τους πράξη πρέπει να λύσουμε άμεσα το θέμα αυτό. Σα ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Καταρχήν, αυτές οι εταιρείε έκδοση καταλόγων επιχειρήσεων δεν χρησιμοποιούν μόνο παραπλανητικές αλλά και απατηλές πρακτικές. Και τέτοιες απάτες βάλλονται κατά τις ίδιες της κοινωνίας. Γιατί με τέτοιες ε, απατηλές πρακτικές οι εταιρείε αυτές προσελκύουν ε, πολίτες και εις βάρος τους ε, κερδοσκοπούν. Αυτό είναι πραγματικά απάτη, δεν είναι απλώς παραπλανητική πρακτική. Και με βάση την οδηγία για συγκριτική παραπλανητική διαφήμιση, οι ε, εταιρείε αυτέ ε, πραγματοποιούν παράνομε δραστηριότητε. Δεν χρειαζόμαστε νέα νομοθεσία, απλώ θα πρέπει να εξασφαλίσουμε εφαρμογή τη ισχύουσα νομοθεσία. Βέβαια, το θέμα είναι διασυνοριακό. Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι μεμονωμένοι έμποροι, δεν μπορούν ε, να προστατεύσουν τον εαυτό τους, ή δεν μπορούν να αναλάβουν την δαπάνη μιας ε, νομικής προσφυγής. Μήπως θα μπορούσε να οργανώσει μια εκστρατεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you, uh, Madam. Ευχαριστώ. Δυόμιση λεπτά, έτσι. Κύριε Επίτροπε, τα τελευταία χρόνια συνάντησα τόσους Ιρλανδούς που ήταν θύματα παραπλανητικών επιχειρηματικών πρακτικών τέτοιων εταιριών. Για παράδειγμα, κάποιο πλήρωσε πάνω από 2.000 ε, ε, ευρώ και αισθάνθηκε ε, άσχημα γιατί έπλεξε το σχολείο και μετά από τύψει δεν ήθελε να επιβαρύνει το σχολείο και πλήρωσε από την τσέπη, από τη τσέπη του ένα φοιτητή. Μία άλλη ηλικιωμένη που είναι σύζυγος ταξιτζή έλαβε το έντυπο με κάποια λάθη, προσπάθησε να τα διορθώσει, αυτό νόμιζε τουλάχιστον, ε, επέστρεψε το έγγραφο και για δύο χρόνια συνέχισε να λαμβάνει απειλητικές επιστολές και μάλιστα είχε τρομοκρατηθεί από τις επιστολές αυτές. Φοβόταν ακόμη και να ανοίξει την, το γράμμα που της έφερνε το χιδρόμος. Τη είπα λοιπόν, μην πληρώσετε ε, δεν μπορούσα να τη πω μην πληρώσετε. Το μόνο που μπορούσα να τη πω ήταν ότι εγώ στη θέση σα δεν θα πλήρωνα. Αυτή ήταν η καλύτερη συμβουλή που θα μπορούσα να δώσω. Υπάρχουν πολλοί άριθμα τέτοια παραδείγματα και όλοι τα γνωρίζουμε. Οι πολίτε περιμένουν ε, προστασία από την κοινοτική νομοθεσία και δεν αντιλαμβάνονται ότι μια κοινοτική νομοθεσία είναι ανίκανη να του προστατεύσει. Υπάρχει μια αμφισημία εδώ και όπως είπα ε, συναντώ πολίτες που πιστεύω ότι θα πρέπει να τη χάνουν προστασία, αλλά δεν μπορώ να του εγγυηθώ τέτοια προστασία. Μία εταιρεία μάλιστα καταδικάστηκε στην Ισπανία και το μόνο που έκανε είναι να μετακομίσει σε άλλη περιοχή και να συνεχίσει ανενόχλητη τι δραστηριότητέ τη. Κάτι άλλο που απασχολεί του πολίτε είναι ότι δεν είναι σίγουροι πώ λειτουργούν τα δικαιωτικά συστήματα άλλων χωρών γιατί μπορεί να αισθάνονται ότι το δικό, η δική τους πατρίδα θα τους προστατεύσει, αλλά δεν είναι βέβαια αν θα τύχουν προστασίες και σε άλλο κράτος. Και πολλές εταιρείες όταν μετακατασταθούν και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμ, ποια θα είναι η θέση των πολιτών, θα τη χάνουν από έξω κοινοτικέ εταιρείε. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να ενημερώσουμε και τις ε, εταιρείε και τους πολίτες. Είπατε ότι είναι επίγον το θέμα, αλλά ε, επίγον θέμα τέτοιο έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι πολίτε πραγματικά δεν καταλαβαίνουν γιατί κολλησιεργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να του προστατεύσει από τέτοιε παραπλανητικές πρακτικέ. Όταν λέμε ότι κάτι είναι κατεπήγον σημαίνει ότι τώρα θα πρέπει να το επιλύσουμε. ο κύριος Στίμψον, για ένα λεπτό. Thank you very much. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, συμφωνώ απόλυτα με την προλαλή σας την κυρία Χάρκιν και εγώ στην εκλογική μου περιφέρεια στη Σκοτία. κυρίως οι ηλικιωμένοι που έχουν ε, πανδοχεία, bed and breakfast, οικογενειακές επιχειρήσεις. Αυτοί είναι που πέφτουν στα δίχτυα τέτοιων κυκλωμάτων και τέτοιων παραπλανητικών πρακτικών. Γιατί βάζουν τις διευθύνσεις τους ε, στον κατάλογο αυτό και τους ζητούν χίλια ευρώ ενώ συνεχίζουν να τους στέλνουν και πολιτικές επιστολές σε περίπτωση που δεν, τους, δεν τα καταβάλουν. Φοβούνται οι ηλικιωμένοι άνθρωποι από τις απειλές αυτών των εταιριών που έχουν διασυνοριακή δραστηριότητα. Γιατί οι εταιρείε αυτές έχουν τα στοιχεία αυτών των ανθρώπων, αλλά και εμείς έχουμε τα στοιχεία των εταιριών. Γιατί να μην, να μην μπορούμε να, τις διώκουμε, αφού έχουμε τις διευθύνσεις τους, το ονοματεπώνυμά τους. Εγώ λέω στους συμπολίτες μου που παραπονιούνται και καταγγέλνουν τέτοια φαινόμενα, στείλτε μου τα στοιχεία των επιχειρήσεων. Όταν το κάνουν, δεν, έχουν, δεν δίνονται συνέχεια στι απειλητικέ επιστολέ. Τώρα από την ομάδα των Πρασίνων για ένα λεπτό επίση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε αυτό το ψήφισμα είναι κάτι που χρειαζόμαστε πραγματικά. Έστω και αν έχουμε την οδηγία του 2006 φαίνεται ότι δεν λειτουργεί ω θα όφιλε. Ε, αυτές ε, οι εταιρείε υπάρχουν έτσι ώστε ε, να δημιουργήσουν προβλήματα στον κόσμο. Και πραγματικά το βρίσκω εξαιρετικά προκλητικό όταν τέτοιου είδους οικονομικές των εταιριών αυτών μπορεί ακόμα και να ε, καταδικάσει ας πούμε οικονομικά ε, μια, έναν οργανισμό κοινοφελή, έναν τοπική αυτοδίκηση κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι ε, κάνουν, πιέζουν με τον χειρότερο τρόπο οι εταιρείε αυτές πραγματικά είναι σαν επιθετικοί καρχαρίες και πρέπει να τις κλείσουμε. Ε, η ομάδα μου καλωσορίζει το ψήφισμα αυτό. Πραγματικά έπρεπε να ε, γίνει και ε, πρέπει να ζητήσει και ο Επίτροπος από τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν σωστά την οδηγία. Την Ευρώπη Ελευθερίας Δημοκρατίας για ένα λεπτό Ε, υπάρχει μια τέτοια εταιρεία, ε, η City Guide ε, Plan, η οποία παρότι έγιναν προσπάθειες να κλείσει τον τελευταίο καιρό, εξακολουθεί και υπάρχει. Κανένας πολίτης τελικά στον οποίο απευθύνεται δεν ξέρει ποια θα είναι ποιο θα είναι το πραγματικό κόστος της υπηρεσίας. Και φαίνεται ότι αυτούς τους αλήτες δεν μπορεί να τους αγγίξει κανένας, ούτε η εθνική νομοθεσία, ούτε η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και εγώ Ακολουθώ από ε, φίλους ε, και ψηφοφόρους να λαμβάνω επιστολές διαμαρτυρίας. Μα δεν είναι δυνατόν να μην μπορούν να προστατευτούν οι συμπολίτε μου από κάτι το οποίο προέρχεται μάλιστα από άλλες χώρες της Ευρώπης. Δεν υπάρχουν εθνικά σύνορα για αυτά τα πράγματα και ακριβώς αυτή η έλλειψη συνόρων όσον αφορά την ε, ε, κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών ε, δίνει την δυνατότητα για παράνομες πράξεις αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστώ. τώρα ερχόμαστε στους άλλους εγγεγραμμένους ομιλητές. Ο κύριος Μπουγιά έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτρο, αγαπητοί συνάδελφοι, θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε την κατάσταση αυτή των παραπλανητικών επιχειρηματικών πρακτικών με τις 400 ε, αναφορές που έχουν στο, δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 5.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή οργανώσεις που έχουν ε, πληγεί και υφίστανται παρενοχλήσεις. 1.000 ευρώ κατά μέσο όρο για μια τριετία από τέτοιου είδους ε, συμβάσεις. Αυτά τα στοιχεία ανακεφαλαιώνουν μόνο εν μέρη τα δεινά των θυμάτων αυτών των παραπλανητικών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν πολύ γρήγορα και τον επιχειρηματικό κίνδυνο και την οικονομική κρίση αλλά και την αβεβαιότητα του μέλλοντος. Πώς θα αποφύγουμε τέτοιες παραπλανητικές ε, ε, πρακτικές για εταιρείε που δεν μπορούν είναι ανήμπορες απέναντι σε τέτοιου είδους ε, πρακτικές. Θα πρέπει να σταματήσουν αυτές οι απάτες γιατί πραγματικά έτσι υπονομεύουμε την οικονομία μας. Γι' αυτό κύριε Επίτροπε θα πρέπει η αναθεώρηση της οδηγίας για τη συγκριτική και παραπλανητική διαφήμιση να επιταχυνθεί λαμβάνοντα υπόψη την, ε, τις εξελίξεις και την εξήτηση που εφαρμόζουν και οι απαταιώνες. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε και, μια μαύρη λίστα των ε, εταιριών αυτών για να τις κατονομάσουμε και να τις ξεμπροστιάσουμε με τη συνεργασία των Εθνικών Αρχών κατά αποτελέμησης απάτης θα μπορούσαμε να έχουμε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό και αποτροπής αλλά και πρόληψης. Τέλος θα πρέπει να επιβάλλουμε κυρώσεις, ποινές, αυστηρές ποινές στους αυτούργους τέτοιων παραπλανητικών πρακτικών. Γιατί οι ποινές και τα πρόστιμα πολλές φορές είναι χαμηλότερα από τα έσοδα αυτών των απαταιώνων. Θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αυστηροί απέναντί τους. Κύριε Γκέμπχαρτ, εκ λόγο για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί και η ανησυχία αυτή είναι και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πάρα πολύ καλό αυτό. Αλλά εδώ και χρόνια περιμένουμε επιτέλου να δραστηριοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να κινηθούν τα πράγματα. Έχουμε την έκθεση του κύριου Μπουζουτήλ στην προηγούμενη θητεία πάντα η Επιτροπή Ιστορικών Υποθέσεων ε, έδινε έμφαση στο θέμα αυτό. Α κάνουμε επιτέλου κάτι για να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται χωρί να του βοηθάμε. Πολλέ μικρέ επιχειρήσει οι οποίε πλήττονται δεν έχουν τα χρηματοοικονομικά μέσα για να αντισταθούν, για να προσπίσουν τα συμφέροντά του. Και την προηγούμενη εβδομάδα πάλι έλαβα μία επιστολή όπου μου ζήτησαν να του πω πώ να αμυνθώ. Δεν έχω χρήματα για δικηγόρο. Νομίζω λοιπόν ότι επιτέλους θα πρέπει να κάνουμε κάτι αποτελεσματικό, να δώσουμε όπλα στα χέρια των πολιτών για να μπορέσουν να ε, σωθούν από αυτή τη μάστιγα. Πολύ, πολύ ακριβής και στον χρόνο. Ε, η κυρία Στήλερ, για, ένα, για ένα, ένα λεπτό παρακαλώ. Ένα λεπτό, κυρία Στήλερ. Thank you, Madam President. the subject... Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε το ε, θέμα αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και επομένως ε, χρειάζεται ε, νομική αντιμετώπιση. Αυτοί είναι αλήτες οι οποίοι δημιουργούν πρόβλημα, απειλούν τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπογράψει κάποια χαρτιά νομίζοντας ότι πρόκειται για δωρεάν υπηρεσία και πραγματικά τους οδηγούν στην απόγνωση. Νομίζω ότι θα πρέπει ο Επίτροπος να σκεφτεί για αυτές τις μικρές επιχειρήσεις πρώτα Πολλοί συνάδελφοι το είπαν ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια γνωρίζουμε την κατάσταση. Πολλά χρόνια διαμαρτυρόμαστε γιατί λαμβάνουμε επιστολές από φίλους και συμπολίτε, και παρόλα αυτά καμία δράση δεν έχει αναλυφθεί. Δράσει χρειάζεται, όχι λόγια, έργα. Ε, γιατί ξέρετε περνάει ο χρόνος, περνάει και ο επόμενος χρόνος και πραγματικά τώρα είναι η ώρα να δράσουμε. Πρόκειται για ε, ε, ανθρώπους που δρούν σε όλη την ε, Ευρώπη. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να τις απειλούν μέχρι όσο δεν αναλαμβάνει η Επιτροπή δράση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λάβει εκατοντάδες ε, ε, αναφορές από μικρές κυρίως επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν πέσει θύματα αυτών των πρακτικών. Ε, πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα προκαλούν πολλές φορές αυτές τις πρακτικές στις μικρές εταιρείες. Πρόκειται για εταιρείες οι οποίες απειλούν και στοχεύουν σε ανθρώπους και θύματα τα οποία ζουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή ε, υπογράφουν κάποιες ε, συμβάσεις με εταιρείε οι οποίες έχουν έδρα σε άλλη ε, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την δικιά τους χώρα. Επίσης οι άνθρωποι αυτοί κάνουν παραπλανητική διαφήμιση και σαφώς παραπλανητικές πρακτικές οι οποίες θα έπρεπε να εμπίπτουν στην σχετική οδηγία. Πρόκειται για συμπολίτε μα οι οποίοι πέφτουν θύματα τέτοιας παραπλανητικής και συγκριτικής ε, διαφήμισης και αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Για ένα λεπτό το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές είναι σαν το νερό. Με το που θα βρουν μία χαραμάδα αμέσως τρυπώνουν μέσα. Και εδώ έχουν βρει δύο χαραμάδες. Η μία χαραμάδα είναι στην οδηγία, η οποία αναφέρθηκε του 2006. Η άλλη λειτουργία, η άλλη χαραμάδα είναι στον κανονισμό που αφορά τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. από τη στιγμή που κύριε επίτροπε έχετε στο πλευρό σας όλες τις πτέρυγες του κοινοβουλίου όλο το κοινοβούλιο πρέπει να δράσετε γρήγορα γιατί ο χρόνος είναι χρήμα και ήδη ανέφεραν οι συνάδελφοι ότι έχουν περάσει τουλάχιστον τρία χρόνια τρία χρόνια κατά τη διάρκεια των οποίων οι άνθρωποι αυτοί οι αλίτες, όπως τους είπαν δικαιολογημένα πάρα πολλοί συνάδελφοι και το προσθέτω και εγώ παραπλανούν συναδέλφους παραπλανούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι ο κορμός της ευρωπαϊκής ένωσης στον οικονομικό τομέα. κάντε κάτι και γρήγορα. ευχαριστώ. ευχαριστώ κυρία ράπτη πολύ ακριβής και στον χρόνο σας. ο κύριος ταραμπέλα για ένα λεπτό. κυρία πρόεδρε κύριε επίτροπε είναι όντω ε, πρωταρχική σημασία να δούμε αν η οδηγία για την συγκρατική και παραπλανητική διαφήμιση έχει όντω σωματωθεί και εφαρμοστεί σωστά στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει αμελητή και ευρυθώ να ασχοληθούμε και με άλλε θεμελιώδει πτυχέ αυτού του ζητήματο, που μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλες μορφές διασυνοριακής απάτης. Καταρχήν θα πρέπει τον των προτέρων να ενημερώνονται οι καταναλωτέ από την Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και τι οργανώσει του. Δεν είναι λογικό να έχουμε όλο και περισσότερου πολίτε που γίνονται θύματα τη απάτης. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα άσκηση λογικής αγωγή από τα θύματα. Περιμένουμε τέτοια ένδικο μέσο εδώ και 20 χρόνια. Σε ό,τι αφορά την ε, μεταρρύθμιση τη. Ε, ε, οδηγίες για, τις εναλλακτικές, ε, για τους εναλλακτικούς διακανονισμούς θα πρέπει σύντομα να προβλέψουμε διατάξει για να διευθετήσουμε το θέμα αυτών των απατών. Περιμένουμε δράση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δικασία Catch the Για ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα υπάρχουν πολλά αιτήματα παρέμβαση. Δεν θα μπορέσουν να πάρουν το λόγο όλοι οι συνάδελφοι, ότι ο χρόνο πιέζει. Μόνο πέντε όσο ήθιστε. Ε, και κυρίω αυτοί που δεν είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν σήμερα το πρωί. Ο κύριο Κέλλη. Ένα λεπτό παρακαλώ, κύριε Κέλλη. Ευχαριστώ. Η κατάσταση είναι ακριβώ όπω μα την περιέγραψαν οι συνάδελφοι. Το ξέρω και από τη δική μου εκλογική περιφέρεια. Εκεί η European City Guide, μια εταιρεία, είχε τέτοιε αθέμητε πρακτικέ απέναντι σε επιχειρήσει. Παρά το γεγονό ε, πω αντιλαμβάνομαι ότι ζητήθηκε ε, από, ε, από ένα δικαστήριο της Καταλωνίας να, να πάυσει τις δραστηριότητες φαίνεται ότι ασκήθηκαν προσφυγές και κατά βελγικών δικαστηρίων και έγινε καταγγελία και στο, στο Βρετανικό Γραφείο Πάταξης της ε, Απάτης. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να λειτουργεί αυτή η εταιρεία. Θα πρέπει να ζητήσουμε τους πολίτες να επαγρυπνούν, να μην πέσουν θύματα αυτών των εταιριών και να θεσπίσουμε για κατάλληλη νομοθεσία ώστε να επιτρέπει στους πολίτες σε περίπτωση που καταγγείλουν μια εταιρεία η οποία θα καταδικαστεί να πάβει τις δραστηριότητές τους και να φυλακίζονται ή να τιμωρούνται οι πέτοι. od podnikatelů neziskových organizací škol charit dokonce i státních institucí které se staly oběťmi podvodů katalogových aktualizace αυτές ε, οι εταιρείε ε, που ασκούν τέτοιες ε, παραπεντικές πρακτικές πολλές φορές προσφέρουν ενημερώσεις για μεγάλα ποσά χρηματικά. Οι δραστηριότητε αυτές είναι διασυνοριακές ή λαμβάνουν χώρα από τρίτες χώρες. Χρειαζόμαστε μια πανευρωπαϊκή λύση. Και θα πρέπει να λάβει δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ κατέθεσα πολλές εναλλακτικέ λύσεις. Θα επαρκούσε αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, καταρτίζει έναν μαύρο κατάλογο, μια μαύρη λίστα με τέτοιες ε, ε, πρακτικές. Χρειαζόμαστε όχι μόνο μια στεναρή ευρωπαϊκή νομοθετική λύση, τη χρειαζόμαστε εδώ και τώρα και ζητώ να εφαρμοστεί η διαδικασία fast track. Έχει το λόγο τώρα για ένα λεπτό παρακαλώ. Eh, Σα ευχαριστώ πολύ. Οι παραπλανητικέ πρακτικέ αυτών των επιχειρήσεων εξακολουθούν να αποτελούν ένα βασικό πρόβλημα. Παρακάμπτουν τον νόμο και ε, βασίζονται στην ε, αμελή εφαρμογή του νομοθεσία. Σε πολλέ περιπτώσει ε, δεν υπάρχει προσφυγή στο δικαστήριο, αλλά σε πολλέ περιπτώσει υπάρχουν και παράλογε δικαστικέ αποφάσει. αλλά οι απαταιώνες ε, βασίζονται στην ε, ελληπή ενημέρωση πολλών νομικών ε, σωμάτων και φυσικά σε πολλές περιπτώσεις μια αμελή εφαρμογή του νόμου. Σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν δεν διώκεται τέτοια συμπεριφορά. Παραδόξως πως σε πολλές περιπτώσεις οι απαταιώνες απολαμβάνουν καλύτερη, νομική καλύτερη... σε νομικής προστασίας από τα θύματα. Πώς λοιπόν σκοπεύετε να επιλύσετε το πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν να επιληθεί το πρόβλημα χωρίς ενεργό δέσμευση των κρατών μελών. Πάμπ, ένα λεπτό όχι παραπάνω. Κύριε Επίτροπε, η ομάδα μας υποστηρίζει την απελευθέρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τη μάστιγα αυτών των εταιριών έκδοσης ε, καταλόγων επιχειρήσεων. Ωστόσο, κύριε Επίτροπε, δικαίως αναφέρατε ότι η Οδηγία 2006-114 προσφέρει μια νομική βάση, ωστόσο κάποια κρατημέλη δεν κατάφεραν να την εφαρμόσουν σωστά. Ελπίζω λοιπόν ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία πλήττονται ιδιαίτερα από το πρόβλημα αυτό να μπορέσουν να καταπολεμήσουν το κακό στη ρίζα του, προκειμένου να επιληφθεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν. Το πρόβλημα είναι, ε, μπορεί να εντοπιστεί σαφώς ορισμένα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η έκδοση καταλόγων επιχειρήσεων είναι ένας πολύ, πολύ χρήσιμη πηγή πληροφόρηση για διάφορες επαγγελματικέ δραστηριότητες και ακριβώς λόγω του κύριου που απολαμβάνουν τη χάνουν και μεγάλης αξιοπιστίε μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών. Οι αθέμητε όμως επιχειρηματικές πρακτικές εταιρείε έκδοσης καταλόγων επιχειρήσεων πλήττουν του πολίτε που προσφεύγουν σε τέτοιε υπηρεσίε. Οι πρακτικές αυτές θα μπορούσαν να σταματήσουν χάρη στην αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας για τη συγκριτική και παραπλανητική διαφήμιση. Δυστυχώς ε, δεν έχουν μεταφέρει όλες οι χώρες ε, την οδηγία αυτή στις ένομες τάξεις τους, γι' αυτό και τα θύματα μένουν ανήμπορα και ανυπεράσπιστα απέναντι σε τέτοιες αθέμητες ε, πρακτικές. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο το συντομότερο δυνατόν και να προβλέψουμε ειδικά μέτρα για να περιοριστεί η εμφάνιση τέτοιων παραπλανητικών πρακτικών. Προσέξει, είχε ζητήσει το, το λόγο από αρκετή ώρα. Ο κύριος Χάφνερ, τελευταίο παρέμβαση. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επιτροπή, αγαπητοί συνάδελφοι, μου φαίνεται ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Όλοι μα και το ακούμε από διάφορε χώρε, γνωρίζουμε τι περιπτώσει αυτέ. Εγώ ξέχω με ένα ολόκληρο ε, φάκελο με τέτοιε περιπτώσει. Και εγώ θα εξαπατώμουν σε πολλέ ε, τέτοιε περιπτώσει. Το πρόβλημα είναι ότι πολλέ φορέ το έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό. Έχουμε την 114 του 2006, το 2008 το συζητήσαμε στην Επιτροπή Αναφορών, το συζητήσαμε στην Ολομέλεια. Το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται και έχει διωγγωθεί μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Ότιγκερ, άκουσα αυτά που είπατε στην αρχή έχω την εντύπωση ότι το πρόβλημα έχει φτάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένα νέο επίτροπος ίσω να έχει μια νέα δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί. Να σα παρακαλέσω να πάρετε στα σοβαρά το πρόβλημα. Μπορεί να φαίνεται μικρό σε έκταση, αλλά οικονομικός πώ είναι πολύ μεγάλο αφορά κυρίω τι μικρέ και με, επιχειρήσει επιχειρήσεις, ε, την ραχοκοκαλιά τη οικονομία μα. Αν δεν καταφέρουμε σε όλα τα κράτη-μέλη να επιλύσουμε τα προβλήματα αυτά, να εφαρμοστεί ενιαία η οδηγία, τότε θα είναι όλο και πιο μεγάλη η ζημιά. Πολύ τελείωσαν οι παραβάσει των συναδέλφων και την ε, ε, ε, συζήτηση θα κλείσει ο Επίτροπος, ο κ. Σέτιγκερ. You have the floor, Mr. Commissioner. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτέ, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για το εύρος και την ομοφωνία στις τάσεις σας και τις ε, τοποθετήσεις σας και για την δέσμευσή σα. Και θα τα αναφέρω όλα αυτά στη συνάδελφο Ρέντινγκ. Και μέχρι τέλη του χρόνου θα συμπεριλάβει τι απόψει σα αυτέ στην σχετική ανακοίνωση. σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας. Καταρχάς διαπιστώνουμε ότι η οδηγία του 2006 έχει εφαρμοστεί στα κράτη-μέλη. Άρα δεν είναι πρόβλημα εφαρμογής μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Αλλά κατά πρώτον, σε διασυνοριακές περιπτώσεις, λόγω της ελλειπούς συνεργασίας των αρχών των κρατών μελών, πολλές περιπτώσεις παρουσιάζονται όπου δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία και δεν υπάρχει σχετική δίωξη. Κατά δεύτερον, συχνά ε, το θέμα είναι η ποινική εφαρμογή. Αυτό το ποινικό σκέλος είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και σε θέματα δίωξης και σε θέματα εφαρμογής από τις ε, εθνικές αρχές, από τις αγγελίες, από τα δικαστηρία. Κατά τρίτον, για να περάσουμε στον πυρήνα της υπόθεσης, η οδηγία του 2006 περιλαμβάνει τις ε, παραπλανητικές ε, πρακτικές αλλά μόνο τις ε, πρακτικές, ε, τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτών. Όχι τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ ε, επιχειρήσεων. Δηλαδή, καταρχάς, αναφέρεται και προστατεύει τον ιδιώτη από τέτοιες παραπλανητικές πρακτικές. Δεν προστατεύει τον πολίτη ως ανεξάρτητο επαγγελματία, ως έμπορο, ως επιχείρηση, ως μικρομεσαία επιχείρηση έναντι των παραπλανητικών αυτών επιχειρήσεων. Ωστόσο, ακριβώς αυτό το στοιχείο διεύρυνσης του εύρους εφαρμογής της οδηγίας και για να συμπεριληφθούν και οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων, αυτό το θέμα στην νομοθετική διαδικασία ήταν κάτι το οποίο δεν ήθελαν τότε τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, τότε ήταν πολύ συνεβητή η επιλογή. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, περιοριστήκαμε στις σχέσεις μεταξύ απαταιώνων και πολιτών και όχι μεταξύ απαταιώνων και μικρών επιχειρήσεων. Άρα αυτό το οποίο καταγγέλουμε τώρα πλέον στην πράξη τότε ήταν ευρωπαϊκή ρύθμιση και ήταν κάτι το οποίο δεν θέλαμε. Η οδηγία τότε αποτελούσε φιλόδοξο ευρωπαϊκό έργο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχούσε ότι δεν θα καταφέρναμε να πετύχουμε καθόλου τίποτα, ούτε καν αυτή την οδηγία. Αν είχαμε επιμείνει στην στάση μας τότε, ενδεχομένως και υπό το φως των συγκεκριμένων παραδειγμάτων που μας έχετε αναφέρει και υπό το φως των ε, ε, ερευνών της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ενδεχομένω λοιπόν να είναι δυνατόν η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή της οδηγία για να συμπεριλάβει και τις επιχειρήσεις. Τέλος, να πούμε ότι υπάρχουν κράτη-μέλη όπου οι απάτες κατά των πολιτών ε, ρυθμίζονται ικανοποιητικά, όπως για παράδειγμα στο Βέλγιο, στην Αυστρία. Υπάρχουν άλλα κράτη-μέλη, έχετε αναφέρει κάποια παραδείγματα, όπου δεν έχουν ρυθμιστεί όλα αυτά με ικανοποιητικό τρόπο στο εθνικό δίκαιο, στην εθνική νομοθεσία. Να δούμε λοιπόν αν αυτά τα κράτη-μέλη είναι διατεθειμένα να προασπίσουν α, μια ευρωπαϊκή, πανευρωπαϊκή τέτοια νομοθεσία για την προστασία του πολίτη. Ε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ε, έλαβα μια πρόταση ψηφίσματος για την ολοκλήρωση αυτής της συζήτησης από την Επιτροπή Αναφορών ε, η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Έληξε εδώ η συζήτηση του θέματος αυτού και ερχόμαστε στο επόμενο